κατέθεσε σύσταση να μην υποβάλει ένσταση κατά πράξη κατά εξουσιοδότηση και αυτή η σύσταση δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2016 και δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις μέσα σε 24 ώρες. Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του κανονισμού θεωρείται λοιπόν ότι η σύσταση αυτή εγκρίθηκε και αύριο λοιπόν δημοσιευτεί με τα σχετικά έγγραφα της ε, συνεδρίασης. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων βάσει του